Ούτε πιστεύω ότι θα πρέπει να συνηγορήσουμε στην επιστροφή αυτών των ανθρώπων σε περιοχές όπου μένεται ο εμφύλιος. Μπορούμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις, αλλά στο τέλος όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος είναι ο τρόπος που προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ από την ομάδα ID η κυρία Ταρδίνο, δύο λεπτά. Έχουμε φτάσει στον ακρότατο βαθμό της δημαγωγίας της αριστεράς. Ανοίξτε τις πόρτες, ελάτε όλοι. Είναι εύκολο να κάνει κανείς τον ευγενικό και το φιλόξενο με τα λιμάνια των άλλων. Θέλετε να δρουν κάποιες οργανώσεις χωρίς κανένα έλεγχο στη Μεσόγειο και θέλετε ότι η δραστηριότητά τους εκφεύγει της εφαρμογής της οδηγίας για την ε, τακτική θα έλεγα μορφή της μετανάστευσης. Εμείς λοιπόν έχουμε καταθέσει μια εναλλακτική πρόταση που θέλει να προστατεύσει πρώτα τα σύνορά μας και μετά τους πολίτες μας. Πρέπει να απαγορεύσουμε τις ε, εκκινήσεις, τις αναχωρήσεις από την Αφρική και πρέπει να ελέγχουμε ε, την προέλευση των ανθρώπων αυτών έτσι ώστε να μπορούμε να δράσουμε στις αιτίε της οικονομικής μετανάστευσης. Μιλάμε πάντα για την ε, λύση του Συμφωνίας της Μάλτα στην αρχή λέγαμε ότι ήταν ε, η λύση για τα πάντα, μετά είπαμε ότι ήταν μια λύση πιλότος πρωτοποριακή και δεν ελέγχουμε όμως έτσι. Δυστυχώς ε, πετύχει για μια ακόμη φορά να ελέγξουμε τις μεταναστευτικές ροές Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να εκτιμούμε σωστά και να αξιολογούμε σωστά την δράση των ιδιοκτικών σκαφών, να δούμε αν πράγματι ασκούν ανθρωπιστική δράση ή είναι απλά κακοπιά στοιχεία. Και θα πρέπει να μην αφήνουν χωρίς λόγο τα σκάφη αυτά να έρχονται στους λιμένες τους ε, χωρίς κανένα έλεγχο θα πρέπει εμείς σε καμία περίπτωση να μην καταστήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες για αυτούς οι οποίοι να μην κατασκήσουν ένα ακόμα κίνητρο για αυτούς που θέλουν παράνομα να έρθουν στην Ευρώπη και μάλιστα πολύ κακοποιοί έρχονται οι οποίοι είναι απλά μεταμφιεσμένοι ουσιαστικά. Συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές ο κύριος Προκατσίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αύριο εμείς δεν θα υποστηρίξουμε την πρόταση αυτή γιατί δεν θέλουμε να είμαστε συνένοχοι αυτών οι οποίοι στην ουσία θέλουν να μην εφαρμόζεται στη Μεσογειακή περιοχή το κράτος δικαίου. Πάρα πολλοί μετανάστες θα φτάσουν ε, θα πέσουν στα χέρια των, ε, ε, των σώματεμπόρων αυτών και γι' αυτό το κόμμα Fratelli d'Italia ε, λέγουν ότι ο μοναδικός τρόπος είναι να απαγορεύσουμε ε, την αναχώρηση των σκαφών αυτών των φουσκωτών από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Είναι η μοναδική λύση. Επαναλαμβάνουμε χωρίς να σταματάμε ότι η διάσωση στη θάλασσα είναι κάτι το οποίο είναι σωστό όταν πρόκειται για κάτι το τυχαίο, κάτι το έκτακτο και όχι κάτι το, οργανωμένο ε, με τη συμμετοχή ε, των σκαφών που ε, υποδέχονται αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Δεν είναι αλληλεγγύη το να δείχνει κανείς ανοιχτές πόρτες στους ανθρώπους αυτούς. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή είναι ένα μανιφέστο σοσιαλιστικής υποκρισίας και γι' αυτό ακριβώς ε, η πολιτική μου ομάδα κατέφεσε ένα εναλλακτικό ψήφισμα. Θέλαμε γραπτός να κάνουμε τις προτάσεις μας και είναι στη διάθεσή σας. Η εκ μέρους της ΓΚΟΕ, ο κύριος Ουρμπαν Κρέσπο. μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάνω από χίλια άτομα πνίγηκαν φέτος στο νεκροταφείο στο οποίο μετατράπηκε η Μεσόγειος. Ε, όταν μπορούμε να διασώσουμε ανθρώπινε ζωέ και δεν το κάνουμε, αυτό είναι ζήτημα ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και όταν τα θεσμικά όργανα δεν κάνουν τίποτα και ποινικοποιούν τις ΜΚΟ, αυτό σημαίνει ότι μετατρέπονται σε συνενόχου. Ε, γιατί ε, το να κλείνουν τα λιμάνια σε, ε, στις σωστικές ε, λέμβους είναι απαράδεκτο. Το να σώζει κανείς ζωές δεν συνιστά ποινικό αδίκημα και η Ευρώπη έχει εκλεονομήσει αυτή την ξενοφοβική στάση από αυτούς τους κυρίους που βρίσκονται εδώ απέναντί μας. Ε, χρειαζόμαστε μια δημόσια ναυτική ασφάλεια στην Ευρώπη. Ε, θα πρέπει να τερματιστεί η παραβίαση των συνόρων. Ε, η Λιβύη δεν είναι ασφαλές ε, λιμάνι θα πρέπει να αλλάξει θα πάνε στην λεγόμενη Λιβιακή ακτοφυλακή. Ε, μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Δεν υπάρχουν ε, ε, ε συγχωροχάρτια όσον αφορά στην παράληψη της διάσωσης ανθρώπινων ζώων. Głos zabierze pan Kostas Papadakis. Półtorej minuty. Bardzo proszę, panie pośle. Ο κύριος Παπαδάκης για τους μη εγγεγραμμένους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τεράστιες ευθύνες της στο υπερελιστικό πόλεμο της Συρίας, όπως και η σύμμαχή της, είναι μέρος του προβλήματος των διωγγούμενων προσφυγικών κυμάτων και όχι της λύσης του. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, το Δουβλίνο και όλε οι ευρωνοσιακέ αποφάσει καταδικάζουν χιλιάδε πρόσφυγε και μετανάστε σε πνιγμό στη Μεσόγειο, σαν το νέο τραγικό ναυάγιο κοντά στην Κο, με νεκρό τρίχρονο παιδί την ίδια ώρα εγκλωβίζονται χιλιάδες άλλοι σε απάνθρωπες συνθήκες στα άθλια hot spots σαν τη μόρια ή τη σάμο τα οποία εδώ και τώρα πρέπει να κλείσουν. η πολιτική της ενίσχυσης των απελάσεων της στρατιωτικοποίησης των συνόρων της καταστολής αποτυπώνεται και στο νέο νομοσχέδιο για το άσυλο της κυβέρνηση νέας δημοκρατίας στην ελλάδα που ανακυκλώνει και οξύνει τα προβλήματα που προκάλεσε η πολιτική της κυβέρνησης του σύριζα. καταδικάζουμε την αλλαγή της ουσίας έννοιας του αιτούντος άσυλου πρόσφυγα τη στοχευμένη επιχείρηση συρρήκνωσης των ήδη τσακισμένων δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών. και οι μεν και οι δε είναι θύματα και δημιουργήματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί επιβάλλει την άμεση μεταφορά του στην υπηρετική ελλάδα σε αξιοπρεπείς δημόσιες δομές φιλοξενίας με μετάβασή του στις χώρες πραγματικού προορισμού του και την υπεράσπιση όλων των δικαιωμάτων των ετούντων άσυλο. οι λαοί λοιπόν σήμερα μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα και με την πάλη του ενάντια σε ευρωπαϊκή ένωση και νάτο να εναντιωθούν στον υπεριαλιστικό πόλεμο να βάλουν εμπόδια στα υπεριαλιστικά σχέδια να απομονώσουν το δηλητήριο του ρατσισμού εθνικισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ο, η κυρία Ετστάντλερ. Ένα μισή λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία ε, Πρόεδρε. Συμφωνούμε επί του πρακτέου. Είναι διεθνές ανθρωπιστικό μας καθήκον να σώζουμε ζωές. Δεύτερον, οι διακινητές, η διακίνηση ανθρώπων είναι από τα χειρότερα εγκλήματα και πρέπει να καταπολεμηθεί με κάθε μέσον. Εμείς μιλάμε για έρευνα και διάσωση εδώ. Στην Αγγλία έγινε καταστροφή ε, ανθρωπιστική. Σε ένα φορτηγό βρέθηκαν 39 ε, πρόσωπα, πτώματα, που ήταν μάλλον ε, πρόσφυγες Επίσης, ε, σε ένα άλλο φορτηγό στη Γερμανία βρέθηκαν 71 νεκροί. Τέτοια περιστατικά μας δείχνουν πόσο αποτρόπαια είναι η διακίνηση ανθρώπων που εκμεταλλεύονται τον κόσμο για να επιτύχουν κέρδη μέσα από το θάνατο των άλλων ανθρώπων. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ τι μηνύματα θα εκπέμψουμε εμείς η έρευνα και η διάσωση στη Μεσόγειο θα πρέπει να ε, εξεταστούν ως προς τα αίτια της. Ε, όσο παραμένουν η Μεσόγειος ένα εισιτήριο για την Ευρώπη θα συνεχίζουν τα προβλήματα. Πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν τις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες να έχουμε καλύτερη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης για να μπορέσουμε έτσι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να εξασφαλίσουμε προοπτικές αυτούς που ε, χρειάζονται. Ο κύριος Μπάρτολο, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Λόμπε Αγγιλάρ γιατί έκανε μια εξαιρετική δουλειά το ψήφισμα αυτό στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με την πολιτική των κεκλεισμένων θυρών. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να θέτουμε σε κίνδυνο στη θάλασσα τη ζωή των ανθρώπων. Πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν μέχρι τώρα είναι ανεπαρκή και απεδείχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο τόξο της Λαμπεδούζα το ναυάγιο. Συνεπώς ε, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους τα κράτη-μέλη και να δώσουν άμεσες και μόνιμες απαντήσεις. Ε, πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν και την έρευνα και διάσωση με κατευθυντήριες γραμμές που να ξεκαθαρίζουν ε, ότι θα πρέπει να βοηθάμε αυτούς οι οποίοι παρέχουν γνήσια ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν μπορούμε να τους απειλούμε ποινικά και θα πρέπει να ξεπεράσουμε εν πάση περιπτώσει τους καταστροφικούς εγωισμούς των κρατών μελών και να μην βρίσκουμε λύσεις ε, μόνο με χώρες σαν τη Λιβύη όπου οι ταλέποροι αυτοί οι άνθρωποι υφίστανται τρομακτική καταστολή και πίεση. Αλλιώς θα είμαστε συνυπεύθυνοι για τις τραγωδίες αυτές και στη Μεσάγειο και όχι μόνο και όποιος δεν λέει τίποτα λέγοντας ότι θα συνεχίσουμε με την συμφωνία με τη Λιβύη που μείωσε τις μετακινήσεις θα πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι δεν μπόρεσαν να διακινδυνεύσουν στη Μεσόγειο ζουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, σε λάγκερ. Το λόγο έχει ο Γιάνν Κρίστοφ για ένα λεπτό. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμε κυρίε και κύριοι, αυτό το οποίο διαδραματίζεται στη Μεσόγειο παραμένει ανθρωπιστική καταστροφή και η διάσωση είναι νομική, ε, νομικό αλλά και ανθρωπιστικό καθήκον. Εμείς ως Ευρωπαίοι έχουμε την ευθύνη να μην κοιτάμε, παρακολουθούμε άπραγοι τους θανάτους στη Μεσόγειο, αλλά να αναλάβουμε δράση. Ε, σήμερα κερδίσαμε μια πλειοψηφία για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων διάσωση. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρο. Αλλά τέσσερις χώρες δεν είναι αρκετές και θα ήθελα να όλες τις χώρες της Ευρώπης να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Το καλύτερο βεβαίως θα ήταν οι άνθρωποι αυτοί να μην επιβαίνουν στα σκάφη. Γι' αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση στους καταβλισμούς, στα στρατόπεδα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε επίσης τις συνθήκες επανεγκατάστασης των πιο αδύναμων και οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν την ευθύνη να συνδράμουν αυτούς τους ανθρώπους. Αναμένω η Κομισιόν να καταστήσει το θέμα αυτό ύψιστη προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τίνε Στρίκ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη θάλασσα κάθε λεπτό μετράει. Είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι θα αφήναμε ε, σε κίνδυνο πνιγμού πολίτες της Ένωσης ε, πλέοντας μέσα σε σχεδίες. Αυτό γίνεται όμως με τους μετανάστες καθημερινά. Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας υποχρεώνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος του Ισουάνκλος να συμμετέχει στην έρευνα και διάσωση διαθέτοντας ε, δυνατότητες επαρκής, ικανότητες στη Μεσόγειο, συντονισμό και αποβίβαση σε ασφαλείς λιμένες. Επειδή η Λιβύη δεν είναι ασφαλής, δεν μπορούμε να ε, οργανώσουμε επιστροφή στην Τρίπολη χωρίς να παραβιάσουμε το διεθνές δίκαιο. Βοηθούμε όμως τους πρόσφυγες να ξεφύγουν από αυτή την κόλαση. Όλα τα κράτη-μέλη γι' αυτό πρέπει να αναλάβουν ευθύνε και να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία πρέπει να ε, προωθείται, όχι να ποινικοποιείται. Οι νέε διευθετήσει θα πρέπει να στηρίζονται σε αυτέ τι αρχέ και πρέπει να είναι ταχείε και μόνιμε. Παρακαλώ, διασφαλίστε τη διάσωση των ζωών των ανθρώπων αυτών και αποβίβαση σε ασφαλεί λιμένε γιατί κάθε λεπτό μετρά. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ζαν Πολ Γκαρό, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση στην ουσία επιτρέπει τη διεύρυνση της μεταναστευτικής πίεσης έτσι ώστε να σωθούν οι ε, μετανάστες ε, από το πνιγμό. Πρέπει να ανοίξουμε όλους τους λιμένες της Ένωσης και να διευκολύνουμε τις εργασίες των ε, ΜΚΙΟ. Στην ουσία να συνεχίσουμε να γινόμεθα πιο ελκυστικοί, να αυξάνουμε τους αριθμούς ε, των ε, μεταναστών που όπως είπε και ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας ε, πέφτουν θύματα του οργανωμένου εγκλήματος με συνενόχους της ΜΚΟ. Αν θέλετε να σώσετε τις ανθρώπινες ζωές και αυτό θέλουμε πρέπει να κάνετε ακριβώς το αντίθετο, να αποκαταστήσετε τα πραγματικά σύνορα στα όρια των Εθνών και της Ένωσης, να διώξετε αυτούς που διευκολύνουν το πέρασμα των δυστυχισμένων μεταναστών, να επιλέγετε τους πραγματικούς ε, δικαιούχους ασύλου και να ενθαρρύνετε τις βοήθειες προς τις χώρες προέλευσης για να αποτρέπουμε τέτοιου είδους δραματικά κύματα, κύματα μετανάστευσης. Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή είναι για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Από την άλλη, οι απαντήσεις είναι σφαλμανμένες γιατί ο αριθμός των ε, θυμάτων ε, αυξήθηκε φέτος σε σχέση με τους περσινούς. Αυτό δεν λέγεται. Η πολιτική μου ομάδα παρουσίασε μία εναλλακτική πρόταση η οποία βασίζεται στις, χώρες, στις αποφάσεις των χωρών μέλη και αφορά την καταπολέμηση των μαφιών που διακινούν τους πρόσφυγες ορθές ε, λύσεις θα ήταν οι εξής. Τι μέτρα θα πρέπει να πάρουμε για να ε, απαλείψουμε αυτό το μοντέλο εμπορίας ανθρώπινων ζώων από τις μαφίες και τις ΜΚΟ που συνεργάζονται με αυτές τις μαφίες γιατί ε, με το, ε, είναι οι χώρες μέλη αυτές οι οποίες έχουν την κυρίαρχη απόφαση κάτω από ποιες ε, προϋποθέσεις υποδέχονται τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπε ο προηγούμενος ομιλητής το 2019 ε, ε, έχουν χάσει τη ζωή τους χίλια ε, άτομα. και υπεύθυνη συνεργασία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί κάνουμε ψηφίσματα καταδικαστικά, αλλά οι πολιτικές δεν αλλάζουν. Αντί να δημιουργηθεί μια, ένα σώμα διάσωσης των ανθρώπινων ζώων, η ε, παρέμβαση στις ζώνες που βρίσκονται συνδρομής ε, και να, ε, ε, σε, ε, όλοι ενέχονται σε μαφίες που προχωρούν στην εμπορία ανθρώπινων ζώων. Ε, υπάρχουν ε, πολυάριθμα περιστατικά πνιγμών και στις ακτές του Μαρόκο. Και θα ήθελα να κλείσω με το εξή. Το διεθνέ Δίκαιο μα υποχρεώνει να διασώσουμε ζωέ. Ελπίζω ότι, αναμένω ότι στην περίπτωση που δεν γίνεται αυτό, θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ κύριος Παλάς Χιτβέγγι, λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή, αυτό το ψήφισμα στηρίζεται σε μια σοβαρή παρανόηση. Η υπέρμαχοί του ισχυρίζεται ότι ο στόχος είναι η διάσωση ζωών, αλλά στην πραγματικότητα η έγκρισή του στέλνει, θα στέλνει το λάθος μήνυμα και θα οδηγούσε σε πιο τραγικά συμβάντα επειδή είναι σαφής πρόσκληση όπως είναι τώρα προς εκατομμύρια ανθρώπους στην Αφρική. Αν ε, ε, κάνουμε σαν να είμαστε ικανοί και έτοιμοι να καλωσορίσουμε τους πάντες στην Ευρώπη, τότε θα έρχονται ακόμη περισσότεροι ρισκάροντας τη ζωή τους. Θα πρέπει να πάμε την βοήθεια εκεί που χρειάζεται, να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του το πρόβλημα. Χρειάζεται να επενδύσουμε στην προστασία των συνόρων, να έχουμε ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, να καταπολεμήσουμε τα κυκλώματα διακίνηση ώστε να μην φεύγουν καταρχήν από τις χώρες τους οι άνθρωποι αυτοί. Ο καλύτερος τρόπος να αποφεύγουμε τους πνιγμούς στη Μεσόγειο είναι να κάνουμε κάθε πολιτική προσπάθεια ώστε οι διακινητέ και τα σκάφη του να μην φεύγουν ποτέ από την ακτή της Αφρικής. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να εμπλέκομαι μη κυβερνητικέ οργανώσεις με ασαφείς δυνατότητε και παρελθόν σε επιχειρήσεις. Ε, είναι τελείως απαράδεκτο να ε, ενθαρρύνουμε τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις να μην ε, τηρούν τους κανόνες και να παραβιάζουν την νομοθεσία. Τα πλοία τους δεν θα πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλουμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές θα πρέπει να ξαναεισαγάγουμε τον έλεγχο των συνόρων και να βοηθήσουμε τις τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στα πλαίσια της ε, γαλάζιας κάρτας ο κύριος Μπιουτικόφερ θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Συμφωνείτε? Κύριε, ο κύριος Μπιουτικόφερ θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Ε, πρόκειται για τη διαδικασία με την γαλάζια κάρτα. Ο κύριος Μπιουτικόφερ θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Συμφωνείτε? Ναι. ναι. Ορίστε λοιπόν, ε, μισό λεπτό κύριε Μπιουτικόφερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις στον συνάδελφο. Πρώτον, είστε βέβαιος ότι ανήκετε στο ΕΛΚ και όχι στο ID. Δεύτερον, αυτά που είπατε είναι χριστιανικά, προσεγγίζουν έστω κατά διάνοια το χριστιανισμό. Η απάντηση τώρα από τον κύριο Χιντβέγγι. Ε, Έτσι κι αλλιώ ε, τέτοιε συζητήσει τι έχουμε κάνει στι πολιτικέ μα ομάδε και ο καθένα λέει ελεύθερα την άποψή του. Δεύτερον, αναφερθήκατε στο χριστιανισμό. Ένα πράγμα να σα πω. Ότι χριστιανισμό σημαίνει υπευθυνότητα. Συνεπώς λοιπόν η Ευρώπη σε σχέση με μετανάστευση είναι ανεύθυνη. Στέλνει τα λάθος μηνύματα στους ανθρώπους αυτούς. Τους λέει ελάτε όλοι, δεν υπάρχουν όρια. Και μετά από λίγο καιρό τους λέμε «Α, κατά λάθο σας δεχθήκαμε, πρέπει να φύγετε». Αυτό είναι ανευθυνότητα. Η υπεύθυνη αντιμετώπιση, η υπεύθυνη στάση είναι να είναι κανείς ρεαλιστής, να δίδει βοήθεια τοπικά στις χώρες που ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστώ. Χαβιέ Μορένο Σάντσες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την προσπάθεια την οποία έκανε που αναφέρεται στα απαραίτητα και κατεπήγοντα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε για να σταματήσουν οι πνιγμοί στη Μεσόγειο. Αυτή είναι η, προσ... προτεραιότητα. Η συμφωνία της Μάλτα είναι ένα θετικό βήμα αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται ανεπαρκές. Θα πρέπει να περάσουμε από τη συνεργασία ανάμεσα σε ορισμένες χώρες σε μια πραγματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατεπήγοντα μέτρα θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και τα παιδιά που πολλές φορές τα παιδιά είναι μη συνοδευόμενα και αντιμετωπίζουν τεράστιους κινδύνους κατά τη διάρκεια της πορείας τους. Ε, χιλιάδες τώρα άνθρωποι ζουν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες ε, στη, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Λιβύης και ανήλικοι Πρέπει λοιπόν να απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να εκενωθούν αυτές ε, οι μονάδες και θα ήθελα να θυμίσω επίσης ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν είναι αριθμοί. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν είναι στατιστικές. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες έχουν μια ιστορία, έχουν μια ζωή, έχουν ένα παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Μαϊτέ Παγαζαοβτουντούα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ δεν αγαπώ την δημαγωγία και σε αυτό το κοινοβούλιο πολλές φορές παρασυρώμεθα ενώ θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή πολιτική ε, στον τομέα του ασύλου και να τελειώνουμε με την κρίση την οποία βιώνουμε. Νομίζω ότι η ανθρώπινη ζωή και σε νομικό επίπεδο είναι θα έλεγα ένα αγαθό το οποίο θα πρέπει να διασώσουμε και από την δράση των ε, σωματεμπόρων και του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη οργάνωση και αστυνόμευση της περιοχής αυτής και νομίζω ότι δεν έχει νόημα τώρα το να μιλάμε με δημαγωγία για ένα τέτοιο πρόβλημα. Θα πρέπει το Συμβούλιο επιτέλους να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Είναι σαφές αυτό που έχουν πει μέχρι τώρα το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε επίσης και τι συμβαίνει στη Λιβύη και δεν μπορούμε να είμαστε απλοί μάρτυρες της συστηματικής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Ευχαριστώ πολύ. Η Κούνκε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κάθε φορά που χάνεται μια ζωή στη Μεσόγειο, αυτό γίνεται γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να αναλάβει δράση. Πνίγομαι από την οργή εγώ. Η έλλειψη αυτή ανθρωπισμού είναι ε, κάτι το οποίο είναι ντροπιαστικό και είναι κάτι το οποίο απάδει στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση συστηματικά και προληπτικά να αναλάβει πλήρως τις ε, έρευνες ε, και την διάσωση στην Μεσόγειο σε συνεργασία πρέπει όλοι να προλαμβάνουμε αυτές τις ε, καταστάσεις, όλοι να ανταλλάσσουν πληροφορίες για σκάφη εν κινδύνο, έτσι ώστε να μπορούν να αναλαμβάνονται οι σωστές δράσεις και κάθε ένας από αυτούς που διασώζονται να μεταφέρεται σε ένα ασφαλή τόπο σύμφωνα με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ. Ο Τόμ Βαντεντρίσε, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, ποιος παραβια... όποιος παραβιάζει τον νόμο τιμωρείται. Έτσι προστατεύουμε τους πολίτες, έτσι εμπιστεύονται το κράτος δικαίου οι πολίτες και αυτό αρνείται να κάνει η πολιτική ελίτ. Αντί να προστατεύει τα σύνορά μας, τους νόμιμους τους μετανάστες που παραβιάζουν ε, το νόμο παίρνουν άδεια παραμονής και κάποιοι εδώ είναι υπέρ των ΜΚΟ που ε, προωθούν την παράνομη μετανάστευση. Αυτή είναι παράνομη. Τι ανθρωπισμός είναι αυτός ε, όταν κρατάμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο διακίνησης ανθρώπων. Πόσο ανθρωπιστικό είναι να ε, βάζουμε τους πολίτες μας ε, να νιώθουν θύματα ε, παρανόμων που διαπράττουν αδικήματα. Δεν πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες κλείνοντας τα σύνορα, προλαμβάνοντας τα μοντέλα διακίνησης για να προστατεύσουμε τους πολίτες. Αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς. Ευχαριστώ η κυρία Βυσνιεύσκα ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να σώζουμε ανθρώπινες ζωές, αλλά οι επιχειρήσεις διάσωσης στην Μεσόγειο συχνά ε, γίνονται ε, αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους διακινητές. Πρόκειται για μια κοινική επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο. Ε, δέκα δις έχουν δοθεί για αυτές τις δράσεις. Η Frontex βέβαια δεν έχει την διάσωση ως βασικό της έργο. Βασικό είναι να μην αφήνει να μπαίνουν παράνομοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ε, έτσι λειτουργούν τα πράγματα χωρίς έλεγχο, χωρίς να ελέγχεται το παρελθόν αυτών των ανθρώπων. Οι επιχειρήσεις διάσωσης δεν πρέπει να είναι ο κανόνας, αλλά η εξαίρεση και γι' αυτό κυρίως θα πρέπει να αναλάβουμε δράση στη στεριά. Όταν ε, εγκρίνουμε μηχανισμό κατανομής, αυτή η κοινική επιχείρηση ε, θα ε, εγκριθεί από εμάς. Πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε ένα ψήφισμα που θα καταπολεμεί τους διακινητές και έχουμε και σχέδιο για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην Αφρική. Έτσι θέλουμε να σταματήσουμε την παράνομη μετανάστευση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μίρια Μντάλη, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως υπογράμμισαν άλλοι συνάδελφοι, η απώλεια ζωών στη Μεσόγειο συνεχίστηκε για πολλά χρόνια. Κι όμως σήμερα ακόμη δεν έχουμε αποτελεσματικό μηχανισμό αλληλεγγύης για τη μετανάστευση. Για κάποια κράτη-μέλη τα προβλήματα των νοτίων χωρών δεν αποτελούν αντικείμενο ανησυχίας. Όμως δεν πρέπει να σταματήσει το έργο μας για να διασφαλίσουμε αξιόπιστη και μόνιμη προσέγγιση στην έρευνα και τη διάσωση που θα αντικαταστήσει τις λύσεις ad hoc που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα ε, δεδομένης της κοινή δήλωση μόνο μεταξύ τεσσάρων χωρών, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Μάλτα, μετά την Υπουργική Σύνοδο στη Μάλτα, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία προβλέψιμου μηχανισμού αλληλεγγύης αλλά μόνο τέσσερα είναι τα κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο θα πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο και να προωθήσει ένα μηχανισμό ίσης κατανομής αυτών που διασώθηκαν στη θάλασσα. Μια προσέγγιση που θα δίνει μεγάλη σημασία στην αρχή της μία ε, παραπρόθεση, αλλά διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες έρευνα και διάσωσης θα τηρούνται και δεν θα γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευση. Τέλος, μια κοινή ενωσιακή απάντηση από όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι η προτιμόμενη λύση. Αλλά αν δεν γίνεται αυτό, ε, δεν μπορούμε να καθόμαστε και να μην πράττουμε τίποτε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χοκ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, μιλάμε μια μέρα όπου, που είναι μαύρη γιατί 39 ε, άνθρωποι ε, μεταξύ αυτών και ένα παιδί ε, βρέθηκαν ε, νεκροί στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι... Και οι εμπειρίες τους διανύει τρεις φάσεις. Καταστροφές στην πατρίδα τους, διέλευση μέσω αφρικανικών χωρών και τέλος αντιμετώπιση των ε, κινδύνων στη Μεσόγειο ακριβώς επειδή δεν έχουν καμία άλλη επιλογή και ε, ορισμένοι από αυτούς ε, γίνονται θύματα και πέφτουν στο έλεος των διακινητών. υπάρχουν ασυνόδευτα παιδιά. Δεν θα έπρεπε να ακούμε σε εκείνου που είναι αντίθετοι προς τη διάσωση. Είναι κατεπίγουσα ανάγκη διάσωση των ανθρώπινων ζώων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, για ένα λεπτό, ο κύριος Ουρτασούν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αύριο το Κοινοβούλιο θα αποστείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή επιχειρήση διάσωση στην ε, Μεσόγειο. Ε, το έχουμε διατυπώσει κατ' επανάληψη και δεν υπάρχει καμία απάντηση από τα θεσμικά όργανα. Εγώ θα ήθελα να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξή. Σα ζητήσαμε να διατυπώσετε συστάσει προ τι χώρε μέλη προκειμένου να ποιηθεί η συνδρομή εκ μέρου των ΜΚΟ. Και από το Συμβούλιο ζητώ να ζητήσει από τις διάφορες χώρες μέλη να σέβονται τι τις υποχρεώσεις όσον αφορά τη διάσωση στη Μεσόγειο, όχι με παθητικό τρόπο, αλλά να αναλάβουν ενεργά μέτρα για την ε, ε, διάσωση. Έχουμε το Δουβλίνο μπλοκαρισμένο. Ωστόσο υπάρχουν τέσσερις ε, χώρες οι οποίες άρχισαν να αναλαμβάνουν την ευθύνη της. Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα. Θα πρέπει ο μηχανισμός αυτός να διευρυνθεί με περισσότερες χώρες προκειμένου να υποστηριχθεί και να εξελιχθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φέστε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο μικρός αριθμός των βουλευτών εδώ δείχνει ότι δεν τους ενδιαφέρει και πολύ το θέμα έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο. Κατ' εξαίρεση οι βουλευτές έχουν δίκιο, γιατί ενώ στη Βόρεια Συρία ε, πεθαίνουν καθημερινά περισσότεροι άνθρωποι ε, από ό,τι στη Μεσόγειο, από έναν άνθρωπο ο οποίος επί δεκαετίες υποστηρίχθηκε από την Ένωση και από την αριστερά και αντιμετωπίστηκε ως εταίρος. Ε, ενώ ήταν σαφές ότι η Τουρκία ε, μετατρέπεται σε κράτος Ισλαμιστικό. Ε, σύντομα θα υπάρξει κύμα προσφύγων από τη Συρία και τις κουρδικές περιοχές. Αντί να επικεντρωθούμε εκεί, πώς θα δημιουργήσουμε ε, προστασία συνόρων και πώς θα αντιμετωπίσουμε τον Δογάν, μιλάμε για την ευθύνη μας για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που κάνουν έρευνα και διάσωση ενώ στην πραγματικότητα διακινούν. Τα πραγματικά προβλήματα δεν είναι πια στη Μεσόγειο. Σταματήστε λοιπόν τα μέτρα έρευνας και διάσωσης, σταματήστε τις παράνομες ΜΚΟ και τις εγκληματικές τους δραστηριότητες και σταματήστε τον εκτοπισμό και την καταστροφή των Κούρδων. Ευχαριστώ. Ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία ε, Πρόεδρε. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, η ροή των ε, μεταναστών έπεσε, μειώθηκε κατά 32% σε σχέση με πέρσι και ο αριθμός των θανάτων στην Μεσόγειο μειώθηκε κατά 42%. Γιατί, ξέρετε, είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής Σαλβίνη, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί για έρευνα, η αύξηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωση στη Μεσόγειο και να γίνουν οι κανόνες πιο ευέλικτοι. Η μόνη εξήγηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει με τη βοήθεια των ΜΚΟ να προωθήσει τη μετανάστευση. Η μαζική μετανάστευση ε, μακροπρόθεσμα κατε, ε, ζημίωσε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις που ε, συνάδουν με τα ευρωπαϊκά ε, συμφέροντα. Θα πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα και να ε, περιθάλψουμε τους πρόσφυγες στις χώρες τους. Ευχαριστώ, κυρία Γκυγιόμ. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τον προηγούμενο Ιούλιο το Συμβούλιο μας είπε ότι ο στόχος είναι ε, η διάσωση των ανθρώπινων ζωών. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη απόσταση με την πραγματικότητα. Η Μεσόγειος γίνεται όλο και πιο φωνική και ε, θυμούμαστε ε, πόσο κατεπίγουσα είναι η ανάγκη να υπάρξει μια επαρκής νομοθεσία σε σχέση με τις αποβιβάσεις των μεταναστών. το επιθυμήσαμε κατά επανάληψη αλλά τίποτα δεν άλλαξε. Ε, θα πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική επιχείρηση διάσωση των ανθρώπινων ζώων, προκειμένου να υπάρξει συντονισμό στου διάφορου ευρωπαϊκού λιμένε. Όσο δεν θα υπάρξει αυτό ο μηχανισμό, θα ε, συνεχίσουν να λειτουργούν οι ΜΚΟ. Γι' αυτό θα πρέπει να τερματιστεί η ποινικοποίηση αυτών των ανθρώπων που υποστηρίζουν του πνιγμένου. Η Κομισιόν εκπώνησε μια οδηγία για την διευκόλυνση της διάσωσης ε, στην προσπάθεια να εξελιχθεί σε μια οδηγία για τη διάσωση των ανθρώπινων ζώων. Ευχαριστούμε. Κυρία Βάουτσμανς. Nu kan ik echt starten. Goedenavond, eh, ε, καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Ένας ε, Βρετανός ποιητής είπε ότι κανείς δεν θα έπρεπε να βάλει ένα παιδί μέσα σε ένα σκάφος εκτός αν ε, οι θάλασσες είναι πιο ασφαλείς από την ξηρά. Αυτό δείχνει ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι θάλασσες δεν είναι ασφαλείς. Ε, από το 2015 έχουν πεθάνει πάρα πολλοί άνθρωποι στη Μεσόγειο και οι αριθμοί αυτοί αυξάνουν γιατί οι χώρες μέλη δίνουν μεγαλοσχήμονες ε, σχέσεις αλλά δεν ε, εφαρμόζονται τίποτα στην πράξη. Πολλές χώρες ποινικοποιούν τις ΜΚΟ επειδή διασώζουν ανθρώπινες ζωές. Ε, πρόκειται για μια πλήρη αντιστροφή των ανθρώπινων ζώων αυτό θα μπορούσαμε να το περιμένουμε από τον Τραμπ ή τον Πούτιν, αλλά εμείς δεν θα έπρεπε να αφήσουμε κανέναν να πνιγεί, αναλαμβάνοντας την ευθύνη μας. Γι' αυτό προσωπική μου παράκληση προς τον κύριο Επίτροπο να ε, διατυπωθεί μια ουσιαστική ευρωπαϊκή πολιτική, ούτως ώστε να μην διευκολύνουμε το έργο των διακινητών. Η κυρία Χούτα Σάιρ. Ε, κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, δείχνει τεράστιες ε, αδυναμίες όσον αφορά τα ανοιχτά της σύνορα τα οποία προσελκύουν πολλούς ανθρώπους από τις χώρες της Ποσαχάριας Αφρικής που επιθυμούν να έχουν μια καλύτερη ζωή. Η, Ευρωπα... η Ευρώπη δεν μπορεί να υποδεχθεί εκατομμύρια Αφρικανούς. Η Ευρώπη ανήκει στους Ευρωπαίους. Η ευρωπαϊκή πολιτική δεν θα πρέπει να μιλούν κατε... χρόνο, ένα χρόνο μετά τον άλλον για την επαναγκατάσταση των ε, προσφύγων. Η Ευρώπη ως ε, σύνολο θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα. Ε, θα πρέπει να συζητούμε το πώς αντιμετωπίζουμε τα εξωτερικά μας σύνορα της Ευρώπης. Το καθήκον μας είναι να διαφυλάξουμε την ευημερία και την ασφάλεια του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ένα λεπτό, η κυρία Ινσίρ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν κολλήσει στις διαπραγματεύσεις για την μελλοντική μεταναστευτική πολιτική. Πνίγεται ο κόσμος στη Μεσόγειο. Αυτό είναι η αλήθεια. Η αντίδραση ορισμένων είναι να ποινικοποιήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που σώζουν ζωές. Ένα σημαντικό κομμάτι του ψηφίσματος που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη είναι να ζητά, ε, ζητεί κατευθυντήριες γραμμές από την Κομισιόν για ε, να, να είναι σαφές ότι η ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς κέρδος δεν είναι παράνομη. Η ευθύνη είναι των κρατών μελών, αλλά λίγες χώρες αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη. Η Συμφωνία της Μάλτας προσπάθησε να κάνει μια κατανομή των ανθρώπων. Αυτό το χαιρετίζουμε. Αλλά πρέπει να βρεθεί μια μόνιμη, μακροπρόθεσμη λύση που θα διασφαλίζει ότι όλοι θα αναλαμβάνουν ευθύνη για ε, μια πολιτική μετανάστευση της Ένωσης που θα είναι σωστή και θα αναλαμβάνουν ε, όλη την ευθύνη των προσφύγων. Και εκείνοι που ε, υπεκφεύγουν λένε ότι προσπαθούν να βοηθήσουν επιτόπου τον κόσμο. Αλλά ε, θέλουν μόνο να αποφύγουν να έρθουν ε, θέλουν να αποφύγουν να έρθουν στην Ευρώπη αυτοί οι άνθρωποι. Ε, κυρία Μπιτζότου. Η συμφωνία της ε, Μάλτα είναι εις βάρος της Ιταλίας και δείχνει ακριβώς τις ανοησίες τις οποίες έκανε η κυβέρνηση στην οποία συμμετείχαν ε, ε, τα Cinque Stelle. Και όλα αυτά με, τους, με τα χειροκροτήματα της υπόλοιπης Ευρώπης αλλά δυστυχώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία επιτρέπει χιλιάδες παρανόμους ε, να έρχονται στην Ιταλία. Αγαπητοί γραφειοκράτες ε, της, των Βρυξελών, πρέπει να μάθετε ότι οι Ιταλοί κουράστηκαν από τις ανοησίες σας και από τις υπερβολές και τις καταχρήσεις σας. Εμείς θα κατέβουμε στα οδοφράγματα για να υπερασπιστούμε τη γη μας και το λαό μας. Δεν θα καταστήσουμε την Ιταλία σε στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, το κοινοβούλιο αυτό θλίβεται για την ε, απώλεια ανθρώπινων ζώων στη Μεσόγειο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Πρώτον, οι πολιτικοί που χρησιμοποιούν όπλα για να επιβάλλουν την ειρήνη στη Βόρεια Αφρική, σύμφωνα με τις δικές τους ιδέες, αλλά δεν προκαλούν τίποτα άλλο παρά χάος. Δεύτερον, εκείνοι που στηρίζουν την μετανάστευση ε, με λάθος οδηγίες ε, και αποφάσεις που δίνουν αθέμητα ε, πλεονεκτήματα στους ε, μετανάστες, ε, όπως επιδόματα κλπ. Εκείνοι που υποστηρίζουν ανθρώπους όπως η κυρία Ρακέτε, που έκανε επιχείρηση διάσωση στη θάλασσα δίνοντας ελπίδες στον κόσμο ότι θα φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και τέλος οι άνθρωποι που οι ίδιοι οι οποίοι πηγαίνουν στη θάλασσα για να ξεφύγουν χωρίς να αξιολογούν τους κινδύνους. Όλοι είναι υπεύθυνοι. Πάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ε, πάνω από δέκα ζητούν χρόνο, δεν θα μπορέσω να τους δώσω το λόγο, όχι σε όλους. Η κυρία Χολμάιερ, η πρώτη ομιλήτρια. Κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, η συζήτηση δείχνει ότι με το ψήφισμα όπως έχει συνταχθεί μόνο μια μικρή πτυχή του προβλήματος καλύπτεται. Και αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Ε, σίγουρα είμαστε υπέρ της έρευνας και της διάσωσης. Δεν υπάρχει διαφωνία στο δημοκρατικό τόξο. Αλλά το να μιλήσουμε μόνο για αυτές δεν, λύνει το πρόβλημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν στην έρημο της Σαχάρας. Και δεν μιλάμε για αυτήν σπάνια γιατί δεν έρχονται σε εμά, δεν είμαστε μάρτυρες, δεν βλέπουμε εικόνες. Και γι' αυτό η μεγάλη προσοχή μας και το έργο μας θα πρέπει να ε, επικεντρωθεί στις ε, περιοχές της Σαχάρας. Ε, εκεί θα πρέπει να βοηθήσουμε. Βεβαίως η έρευνα και η διάσωση καταξιώνει το έργο της Frontex. Πάρα πολλοί άνθρωποι σώζεται. Αλλά η λύση, αν περιοριστεί εκεί, δυστυχώς δεν είναι λύση. Ο κύριος Σαλίμπα, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, οι υπάρχουσες λύσεις δεν επαρκούν. Είναι προφανές ότι δεν είναι ικανές να αντιμετωπίσουν την παρούσα κρίση. Από τη μία έχουμε τους μετανάστες, γυναίκες και παιδιά να εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους ε, στην ε, ε, Μεσόγειο θάλασσα. Από την άλλη έχουμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι λόγω ακριβώς της αδράνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης νότιες συνοριακές με την περιοχή χώρες ε, βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όπως η Μάλτα. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε να είμαστε αδρανείς. Αυτό ανησυχεί τους συμπολίτε μας και ε, θα αυξηθούν οι βίες ε, ιδεολογίες θα πρέπει να υπάρξει λογική και αλληλεγγύη για μια κοινή λύση. Η κυρία Γιοφέβα για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί επιτέλους ε, η τραγωδία στη Μεσόγειο. Δεν πρέπει όμως να μένουμε στα λόγια, πρέπει να κάνουμε τα συγκεκριμένα βήματα που απαιτούνται. Και ακριβώς αυτό προτείνει το ψήφισμα. Καλύτερος συντονισμός ε, για τη διάσωση ε, και την αποβίβαση των μεταναστών στη Μάλτα και σε άλλες χώρες. Πάνω από 19.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πέρυσι. Αυτό είναι τρομακτικό. Καταλαβαίνω ότι το θέμα αυτό άπτεται και προβλημάτων ασφαλείας, αλλά η αλληλεγγύη με την ασφάλεια μπορούν να συμβαδίσουν. Τα κράτη-μέλη μπορούν να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους και να βρουν πράγματι καταφύγιο στην Ευρώπη αυτοί οι οποίοι έχουν ανάγκη. Ο κύριος Μπεζίνσκι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καταρχήν θα ήθελα να σας αναφέρω ένα παράθωμα. Όποιος σώζει μια ανθρώπινη ζωή, διασώζει ολόκληρο τον κόσμο. Και θα ήθελα να αφαιρθώ στη δική μου εμπειρία υπήρξα, διατέλεσα ναυτικός. Εάν ε, κανείς βλέπει έναν άνθρωπο στη θάλασσα πρέπει να τον βοηθήσει. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Αλλά ως ε, πολιτικός, ως υπεύθυνο άτομο γνωρίζω ότι ε, παρακολουθούν τη σύντησή μας και εγκληματικές οργανώσεις και επίσης και άνθρωποι που ζουν στην Αφρική. Εγώ ήμουνα υπουργός φρετορικών στην Πολωνία και πριν από δύο χρόνια στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου άκουσα μόνο μία λογική φωνή όταν ο Υπουργός Φρετορικών του Μαρόκο είπε ότι πρόκειται για μία πραγματική εισβολή. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνουμε εδώ ενθαρρύνει αυτούς τους ανθρώπους να μεταβούν από την Αφρική στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, θα μιλήσω ένα... Παρακαλώ να μιλήσετε ένα λεπτό. Ε, Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στα 39 θύματα που βρέθηκαν ε, σε ένα φορτηγό στο Essex μέσω του Βελιού ε, από μια Ιρλανδική επιχείρηση η οποία ήταν καταχωρημένη στην Βουλγαρία. Ε, πρόκειται για ένα τραγικό και πραγματικά σπαρακτικό παράδειγμα του πόσο απελπισμένοι είναι οι άνθρωποι και τι κινδύνους, ε, τι ρίσκα παίρνουν για να έρθουν στην Ευρώπη. Χαιρετίζω αυτούς ε, που προσπαθούν να διασώσουν ανθρώπινους ζωές σύμφωνα με την ηθική και το διεθνές δίκαιο. Αλλά τι κάνει το διεθνές δίκαιο τελικά επαναπροωθεί τους ανθρώπους πίσω ή στη Λιβύη όπου αντιμετωπίζουν καταστροφικές συνθήκες. Χρειάζεται να μεταρρυθμιστεί η συνθήκη, να θεωρηθεί η συνθήκη του Δοβλίνου και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση. Αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να πάψουμε να βομβαρδίζουμε τις χώρες τους ε, παράγοντας συνεχώς ε, πρόσφυγες. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα λεπτό για τον κύριο Πόλτσακ. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε, είδατε πόσοι συνάδελφοι από την ομάδα IDF e έφυγαν χωρίς να περιμένουν καν τη δήλωση του Επιτρόπου. Είναι ντροπή, δεδομένου πόσες αντιρρήσεις εξέφρασαν κατά του ζητήματος και της πολιτικής μας. Είναι απαράδεκτο να πεθαίνουν ε, τόσοι άνθρωποι στη Μεσόγειο. Είναι ντροπή για την Ευρώπη. Από την άλλη, δεν μπορεί η ΜΚΟ να εργάζονται ως θαλάσσια ταξί και να αντικαθιστούν τη Frontex. Αυτό είναι όντως απαράδεκτο. Και οδηγεί σε άλλα προβλήματα, όπως κινδύνους ασφαλείας, στήριξη του οργανωμένου εγκλήματος. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα και έχουν να κάνουν με την αντικατάσταση των κυβερνήσεων από ΜΚΟ. Δεν πρέπει να απόσχουμε από την Μεσόγειο. Ο κύριος Ματσολίνο, ένα λεπτό. Εγώ άκουσα φρικτά πράγματα από πλευρά τη δεξιά. Έχουμε να κάνουμε με μια απλή επιλογή μέσω αυτού του ψηφίσματος πρέπει να διασωθούν οι ανθρώπινες ζωές. Αυτό φυσικά δεν φτάνει από μόνο του. Κανένας δεν λέει ε, στους μετανάστες ελάτε όλοι. Εμείς λέμε απλά να διασώσουμε τις ζωές που είναι σε κίνδυνο. Και ας καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο λείπει, μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Το λέω σαν Ιταλός αναδιανομής των μεταναστών στο ευρωπαϊκό έδαφος. Πρέπει να ξεπεραστεί ο κανονισμός του Δουβλίνου, πρέπει να ενεργοποιηθούν οι νόμιμοι οδοί εισόδου. Αυτά είναι τα πραγματικά όπλα εναντίον των σώματεμπόρων. Νομίζω ότι ε, έχουμε απέναντί μας μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία δεν αποδίδει και ε, πρέπει να προστατεύσουμε τις ζωές αυτές και να μην τις θέσουμε σε κίνδυνο για λίγα ψηφαλάκια. Ο Επίτροπος έχει το λόγο για να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, όπως είπα στην αρχή, το να διασώσουμε τις ζωές πάντα ήταν και θα συνεχίσει να είναι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η ηθικό μας καθήκον το να διασώζουμε ζωές και να προστατεύουμε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να αποφύγουν τον θάνατο και την καταστροφή. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε μια ευρωπαϊκή αποτελεσματική στρατηγική για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Θα πρέπει επίσης να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε τις βασικές αιτίες τις ρίζες από τις οποίες ε, μεγενθύνεται η κρίση αυτή. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τους δουλεμπόρους οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα ευάλωτα χαρακτηριστικά των πληθυσμών αυτών και να διευκολύνουμε τους νόμιμους, ε, τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί μόνη της να το πετύχει, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαστόμεθα με τις χώρες διαμετακόμισης και με τις χώρες προέλευσης. Έτσι, σε συνεργασία και με τις ΜΚΟ, μέσω της κατανομής των ευθυνών, στα πλαίσια ενός πνεύματος διεθνούς συνεργασίας θα πετύχουμε. Όλα αυτά νομίζω θα αντικατοπτριστούν ε, στο νέο πακέτο το οποίο θα παρουσιάσει η Ursula von der Leyen ε, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές προκλήσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ. Η Υπουργό του Περάινεν έχει το λόγο. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, η Φιλανδική Προεδρία γνωρίζει πολύ καλά την τεράστια σημασία της ανθρωπιστικής κατάστασης και βοήθεια στη Μεσόγειο και έχουμε δέσμευση να εργαστούμε σε πιο στέρεη βάση, για μια πιο στέρεη λύση, συνεργαζόμενη με όλους τους εμπλεκομένους. Μια τέτοια διευθέτηση πρέπει να είναι προβλέψιμη σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας για την αποβίβαση ε, που θα επιτρέπει ε, διαδικασία ασύλου σωστή και επιστροφή όπου δει. Είναι σημαντικό να επιτύχουμε γρήγορα. Όμως χρειάζεται λύση που θα καλύπτει όλες τις πτυχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και οι ίδιοι οι μετανάστες δεν αξίζουν ε, ε, αυτή την κατάσταση να μένει ανεπίλητο το πρόβλημα δηλαδή πρέπει να σώζουμε ζωές μιλάμε για ανθρώπους εδώ μιλάμε για πρόσωπα Παράλληλα, συνεχίζομαι προς τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου για να δοθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα στο μέλλον. Παραμένω αισιόδοξη ότι χάρη στις προσπάθειές μας θα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά προς την επίτευξη του στόχου μας. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ ε, πρόεδρε της Επιτροπής Λίμπε. Ε, για την υποστήριξη. Το έργο συνεχίζεται. Ευχαριστούμε κυρία του Ράινεν. Υπάρχουν τέσσερις προτάσεις ψηφίσματος ε, μετά από αυτή τη συζήτηση. Οι, τα, οι τέσσερις προτάσεις θα τεθούν σε ψηφοφορία αύριο. Και προχωρούμε τώρα στην επόμενη συζήτηση η οποία είναι δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Πριν να ανοίξω τη συζήτηση, πρέπει να σα πω ότι αν θέλετε ε, να συμμετέχετε στο Catch the Eye, η γαλάζια κάρτα, ε, έχουμε νέο σύστημα, δηλώνεστε ηλεκτρονικά, οι οδηγίε είναι στο έδρανό σα και με τη γαλάζια κάρτα και με το Catch the Eye. Και μπορεί να γίνει αυτό όχι στο τέλος της συζήτησης, αλλά οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Δηλωθείτε όποτε το επιθυμείτε. Όλοι είναι έτοιμοι, κυρία Υπουργέ, έχετε και πάλι το λόγο. Η κυρία του αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η πρόοδο τη Βόρεια Μακεδονία και τη Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Οδό συζητήθηκε στο Συμβούλιο για αρκετό χρονικό διάστημα. Γνωρίζετε επίσης, και το ξέρω, ότι το Συμβούλιο ακόμα δεν μπόρεσε να φτάσει σε συμφωνία μετά τις συστάσεις της Κομισιόν να ανοίξει τις διαπραγματεύσεις ένταξης με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Εν τω μεταξύ και οι δύο χώρες εργάστηκαν σκληρά για να προχωρήσουν τις μεταρρυθμίσεις τους. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου από τον Ιούνιο μας ε, ε, βοήθησαν μας είπαν ότι θα λαμβάναμε το αργότερο τον Οκτώβριο αποφάσει για τις δύο χώρε. Ως πρόεδρος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων πρέπει να πω ότι είμαι βαθιά απογοητευμένη διότι αποτύχαμε να